αυτές προτάσεις. Η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς έχει στείλει ένα διορθωτικό σημείο μας σύμφωνα με το άρθρο 231 του κανονισμού. Θεωρείται ότι έχει εγκριθεί αυτή η διόρθωση. Εάν εντός 24 ωρών δεν εγερθεί καμία αντίρρηση από ε, μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές που θα ζητούν να ψηφιστεί. Το κείμενο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα ε, της Ολομέλειας και ε, στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα δημοσιευθεί ο τίτλος. επτά ε, προτάσεις θα υπογράψω μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου την Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο